Ε, με την ε, αποτροπή της συγχωρήπανσης. Σκοπός μας είναι να έχουμε όσο πιο πολλούς επιβάτες γίνεται στις συντροτροχές προκειμένου. Σας ευχαριστώ, διακόπτη ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, λέει ο Πρόεδρος, να σας ζητήσω, συνάδελφοι, να μιλάτε λίγο πιο σιγά. Γιατί οι τριμηνείς αντιμετωπίζουν προβλήματα με τόσο γρήγορες ομιλίες. Ο Σαΐτ Ελκαντράουι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγή.